και με αυτές τις προτάσεις να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό αλλά και πιο δίκαιο σύστημα ΦΠΑ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσαν Στις 11.30 αύριο θα γίνει ψηφορία αυτής της έκθεσης και τώρα. Περνούμε στο επόμενο θέμα. Βοήθεια κατεπίγουσα προς την ΑΕΤ. Η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Και σε incorpora rápidamente a su sitio η οποία σπέβδει προς το εδρανό της. Thank you, Mr. Chairman. The Commission is deeply concerned by the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την επιδείνωση τη κατάσταση τη χολέρας στην ΑΕΤ. Ο αριθμό των θυμάτων και των νοσηλευομένων αυξάνεται ραγδαία καθημερινά. Η ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο έχουν φτάσει πλέον τις 20.000 ε, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας συγκεκριμένα. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους. Όμως υπάρχει ο φόβος ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν ε, δεν είναι ακριβή, Είναι πολύ υψηλό το ποσοστό θνησιμότητας και φαίνεται ότι στα νοσηλευτικά κέντρα φτάνουν πολύ αργά οι ασθενείς. Είναι απλή η αγωγή για την χολέρα, όμω η έγκαιρη πρόσβαση στην ε, νοσηλεία είναι κάτι που μπορεί να λύσει πολλέ φορέ το πρόβλημα, να σώσει ζωέ. Και βεβαίω εδώ απαιτούνται και ανθρώπινοι πόροι. Το νοσηλευτικό σύστημα τη ΑΕΤ προφανώ δέχεται υπερβολικέ πιέσει παρά την σοβαρή στήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Η γιατροί χωρί σύνορα ήταν ένα από του πρώτου ιατρικού παράγοντε που ανέλαβε δράση και καλεί όλα τα ιδρύματα και τους, τις καθώ καθώς και τον πρόεδρο της ΑΕΤ να ε, επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Αυτή τη στιγμή πλήττεται ολόκληρη η χώρα. Η επιδημία ε, ραγδαία στο Πόρτο Πρέν στην πρωτεύουσα εξαπλώνεται αλλά και σε διάφορες ε, παραγκουπόλεις και στα προάστια υπάρχει το ίδιο πρόβλημα λόγω του κακού αποχετευτικού συστήματος και της έλλειψης πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Ε, η περίθαλψη λοιπόν των ασθενών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, η σωστή συμπεριφορά υγιεινής καθώς και ιατρική παρακολούθηση είναι θέματα που πρέπει να τα προωθήσουμε ώστε να αντιμετωπιστεί η επιδημία. Η Επιτροπή έχει ενισχύσει την ανθρωπιστική της παρουσία με ε, ε, υπεύθυνου ιατρικούς εμπειρογνώμονες και κινητοποιώντας ένα κονδύλι 12.000 ε, ευρώ, 12 εκατομμυρίων ευρώ, συγγνώμη, για να ενισχύσει την IT. Εδώ η παρακολούθηση και το σύστημα ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναλάβει δράση και έχει συγχρηματοδοτήσει την μεταφορά ιατρική στήριξη που προσέφερε η Γαλλία. Μια άλλη προσφορά τη Αυστρία ήδη έχει περάσει στην ε, πορεία της προς την ΑΕΤ και θα δείτε ότι με την στήριξη των ε, εμπειρογνωμών των 100 μελών ε, άμεσα στην αρχή της εβδομάδας αυτής θα γίνουν περαιτέρω βήματα. Η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχει αναλάβει δράση επίσης για να βελτιώσει την επιδημιολογική επαγρύπνηση στην ΑΕΤ και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε και άλλες μορφές συνεργασίας. Μετά τα πρόσφατα περιστατικά, τα κρούσματα που ε, παρατηρήθηκαν στο ΚΑΠ ε, της ΑΙΤΙΣ, ε, στο κοτήρι της ΑΙΤΙΣ και στο Πόρτο Πράνς βλέπουμε ακριβώς πώς δρούν εκεί οι ανθρωπιστικοί φορείς, ιδίως με την προοπτική των προεδρικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τον, με τον με την κυρία με την Παρόνη Έμος που είναι η δεύτερη γραμματέα των Ηνωμένων υπεύθυνη για το θέμα αυτό και βεβαίω ε, συζητούμε με όλου του εργαζομένου στι ανθρωπιστικέ οργανώσει και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να νοικοδομηθεί. Ε, λόγω τη σοβαρή και ταχύτατη επιδείνωση τη κατάσταση με τη χολέρα, θα πρέπει να ε, έχουμε περαιτέρω συνεισφορά από την πλευρά όλων ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με το νερό, τη διοικητική οργάνωση, την περίθαλψη και την οσυλία το ιατρικό προσωπικό, καθώ και οι εργάτε που μπορούν να εξασφαλίσουν την μεταφορά του νερού, η νοσηλεία, ιατρικό υλικό, εγκαταστάσει, ε, κλίνε, όλα αυτά είναι πράγματα που λείπουν στην ΑΕΤ. Γι' αυτό με τη βοήθεια τη Βελγική Προεδρία και των κρατών μελών θα πρέπει η Επιτροπή να προσφέρει περισσότερη βοήθεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΑΕΤ που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Η ευρωπαϊκή βοήθεια μπορεί να κατευθυνθεί στην ΑΕΤ μέσω της, των μηχανισμών πολιτική προστασία που διαθέτουμε. Επίση, οι εργαζόμενοι στον τομέα των ανθρωπιστικών οργανώσεων πρέπει να ενισχυθούν για να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει στην πράξη. Διότι η κλίμακα, οι διαστάσεις της, κρίση κρίσης δείχνουν ότι χρειάζονται περισσότερε προσπάθειες και περισσότεροι πόροι. Πρέπει να επιταχύνουμε την δυνατότητα αποκρισή μα σε επίγοντα περιστατικά μαζί με του εταίρου μα. Όμω, η δύσκολη καιρή είναι ακόμα μπροστά μα, διότι όπω είπα η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία και καθημερινά. Η σταθερή αλληλεγγύη τη διεθνού κοινότητα προ τον λαό τη ΑΕΤ είναι μια προτεραιότητα ουσιαστική. Γι' αυτό σας καλώ όλους σας να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να ε, ενισχυθεί η βοήθεια των κατών μελών και να αποφύγουμε μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε. Και τώρα περνούμε στους αγορητές των πολιτικών ομάδων και για 1,5 λεπτό για το ΕΛΚ η κυρία Στρίφλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Δαμανάκη, η επιδημία της χολέρας ήδη έχει προκαλέσει 1.200 θανάτους και ε, πάνω από 5.000 άτομα έχουν μολυνθεί. Η κατάσταση στην Αιτή χειροτερεύει από τη μία μέρα στην άλλη και στους επόμενους ε, μήνες η επιδημία μπορεί να πλήξει 400.000 άτομα. Βέβαια χαίρομαι για τις πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αξιολογώ ότι την έκκληση της Επιτρόπου Γεώργεβα προς ε, την ε, ε, τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν σε μηχανήματα για να καθαριστεί το πόσιμο είδωρ η μία από τις πρώτες ενέργειες είναι τα άτομα τα οποία φοβούνται την ασθένεια που είναι άγνωστη στη χώρα και θα πρέπει να πληροφορηθεί ο πληθυσμός για να αποφευθούν εσωτερικές βίες διότι είναι προεκλογικής περίοδος. Αυτή η κρίση τόνισε ακόμη μία φορά την αδυναμία των αρχών της ΑΕΤ και του συστήματος υγείας να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Αιτή, υφίσταται πολλές καταστροφές εδώ και χρόνια. Ο σεισμός απέδειξε την ε, ε, ανικανότητα των τοπικών αρχών. Υπήρχε η πολιτική βούληση να ε, ανοικοδομηθεί διαφορετικά η Αϊτή αλλά εδώ και ένα χρόνο είμαστε απεσιόδοξοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να βοηθήσει για να αντεπεξέλθει και να βγει το χάο η IT. Ευχαριστούμε κύριε Στίβλα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες και για ένα λεπτό έχει το λόγο κυρία Κρέτου. Κύριε Πρόεδρε, αξιολογώ τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αντιδράσει και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε το κράτος να λειτουργήσει σωστά και δεν υπάρχει καν κράτος. Ε, υπάρχουν ε, καταλήματα προσφύγων και δεν είναι δυνατόν ε, να ρυθμιστούν τα ουσιαστικά θέματα. Γι' αυτό και πέθαναν ήδη 1200 άτομα. Δηλαδή η IT χρειάζεται δομές να βοηθήσει τους στοχούς γιατί οι τρεις στους τέσσερις ανθρώπους στην IT ζουν με λιγότερο από δύο δολάρια την ημέρα και τα καταλήματα των προσφύγων ε, του σεισμού επιδεινώνουν την κατάσταση και η έλλειψη ε, μια σταθερής εξουσίας δείχνει ότι ο πληθυσμός μπορεί μόνο να, βοηθήσει, να βοηθηθεί από τον ΟΗΕ που δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και τώρα έχω έχουμε εκλογές και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν θα ρυθμιστούν σωστά. Ευχαριστούμε κυρία Κρέτου για, για την ε, Συμμαχία Φιλελευθέρων Δημοκρατών και το λόγο κύριος Γκέρνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και βέβαια έχουμε αυτές τις μεταβλητές που έχουν ε, βοηθήσει την χολέρα να εξαπλωθεί. Αυτό δεν είναι όμως η απάντηση, είναι μια ε, εξήγηση και σε πρώτη φάση η απάντηση θα πρέπει να είναι η ανθρωπιστική βοήθεια επιτόπου για να μπορέσει να υπάρχει πόσιμο είδωρ και επίσης και να υπάρχει κατάλληλη ε, εκπαίδευση όσον αφορά την υγιεινή γιατί πρόκειται για μια χώρα που θα πρέπει όλοι να ξαναγίνουν από την αρχή οπότε επιβάλλει τώρα να γίνει η ανοικοδόμηση της χώρας μετά από αυτόν τον ε, σεισμό οπότε και θα πρέπει τώρα να έχουμε κάποια υποδομή που θα βοηθήσει και την ατομική αλλά και την συλλογική υγιεινή. Και τολμώ να πιστεύω ότι οκτώ μήνες μετά την διάσκεψη της Νέας Υόρκης για την ασυγκρότηση της χώρας δεν μπορούμε πια να έχουμε καμία δικαιολογία ελλείψης χρημάτων ούτως ώστε να εξηγηθεί η πάρα πολύ μικρή πρόοδος μέχρι σήμερα και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναγνωρίσουν ότι θα πρέπει να παρατηθεί ακόμα η διάρκεια συνεργικής βοήθειας να μην ε, αργούμε τόσο πολύ και να προχωρήσουμε με προσοχή. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρινς και τώρα για τους πρασίνους. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Είδαμε ότι είχαμε μία από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα εκείνη και θα πρέπει να μην χαθεί η μάχη κατά της θεομηνίας, να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Ο κόσμος εκεί να μπορέσει να ξαναχθεί στο μέλλον του και μετά από αυτή την καταστροφή μετά από τόσα εκατομμύρια που επλήγησαν όλη η παγκόσμια κοινότητα ε, τώρα αμαυρώθηκε που δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο έπρεπε και άρα θα πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα από την ΑΕΤ, από αλλού να μπορέσουμε να δώσουμε όλα τα χρήματα που χρειάζονται οπότε και εγώ χαιρετώ το ότι θα δώσει η Κομισιόνα ακόμα 12 εκατομμύρια ευρώ κατά της χολέρας. Θα πρέπει να δοθεί όλη μαζί βοήθεια και όχι σε δόσεις για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική και να εξασφαλίσουμε επίσης το ότι δεν θα σταματήσει η βοήθεια προς τη χώρα αυτή για την ασυγκρότηση κατόπιν του σεισμού γιατί αυτό συνδέεται με την αντιμετώπιση της χολέρας. Δύο ερωτήσεις. Τι έγινε με τα χρήματα τα οποία είχαμε υποσχεθεί. Δόθηκαν, απορροφήθηκαν. Επίσης, τι πιστεύετε για το θέμα των εκλογών. Πρέπει να αναβληθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πράγμα στη χώρα τώρα. Αλλά η ιστορία θα καταγράψει ότι τώρα γίνεται μια νέα αρχή. Και επίση τώρα θα γράψει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε θετικό ρόλο σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κέλλερ. Και τώρα για του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ και για ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν από δύο μήνε ήμουν μαζί με μια αντιπροσωπεία στην ΑΕΤ υπεύθυνη αντιπροσωπεία για τι χώρε, ΑΚΕ και ήταν από τι πιο συγκινητικέ εμπειρίε τη ζωή μου αυτή διότι ήταν πάρα πολλοί οι άνθρωποι που εργάζονται για να βοηθήσουν το λαό της ΑΕΤΗΣ. Και είναι και πολύ περήφανοι οι άνθρωποι της ΑΕΤ. Και αυτό δεν πρέπει να το, παραμε... να το αμελούμε κατά τη διάρκεια της συζήτησή μα. Πάντως ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκαν ότι ήταν πολύ τυχεροί οι Αιτενοί τώρα που δεν είχαν προβλήματα με ασθένειες και καλό σύστημα υγείας. Να λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Η ασθένεια αυτή, η επιδημία, δεν είναι δύσκολο να θεραπευτεί. Όμως βλέπουμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει και βλέπουμε τι προσπάθειες κάνουν οι εργαζόμενοι στι ανθρωπιστικέ οργανώσει Βλέπουμε ότι το σύστημα υγείας βασίζεται στους γιατρούς χωρίς σύνορα και πάρα πολλές άλλες οργανώσεις από όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι σε ό,τι αφορά τι εκλογέ τη ΑΕΤ, σίγουρα δεν είναι καταλληλότερη στιγμή για να γίνουν προεδρικέ εκλογέ στην ΑΕΤ. Όμω μέχρι να υπάρχει πρόεδρο και πρωθυπουργό που θα μπορέσουν να ηγηθούν τη χώρα, η χώρα αυτή δεν θα μπορέσει να προοδεύσει. Είμαι βέβαιο γι' αυτό και συστήνω λοιπόν εδώ η ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τόσο δυνατούς επιτρόπους ε, γυναίκες και άντρες να διασφαλίσει μέσω του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη βοήθεια προς την ΑΕΤ. Ευχαριστούμε για την ε, Ενωμένη Αριστερά η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων, ιδιών τη διάσκεψη των Προέδρων, οι οποίοι δέχτηκαν να γίνει αυτή η συζήτηση για την ΑΕΤ που πρότεινε η δική μα ομάδα. Ήταν ένα θέμα κατεπήγον τον περασμένο Ιανουάριο μετά το σεισμό. Η διεθνή κοινότητα κινητοποιήθηκε ε, σοβαρά για να βοηθήσει την ΑΕΤ. Όμω από τι υποσχέσει και τι βοήθειε που ακούσαμε να γίνονται και να φτάνουν και στη χώρα συγκεκριμένα, από τότε δεν έγιναν πολλά. Το περασμένο Μάρτιο η Βερονιά ε, δεσμεύτηκε να διαθέσει 1 δις 350 εκατομμύρια ευρώ στον λαό της Αιτής ε, για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον, μέλλον όπως είπε. Το περασμένο Ιούλιο, κύριε Επίτροπε, όμως ε, είδαμε να μην έχουν γίνει πολλά. Θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η ανθρωπιστική κατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα που ε, λαμβάνει τέτοιε διαστάσεις η επιδημία τη χολέρα. Η διεθνή κοινότητα λοιπόν τώρα πάλι αρχίζει να συγκινείται. Ήδη έχουμε εκατοντάδε χιλιάδε νεκρούς. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, διότι οι γιατροί μας λένε ότι είναι απλή θεραπεία της ασθένειας, αλλά πρέπει να έχει έγκαιρη αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα, τα ιατρικά προϊόντα πρώτης ανάγκη, δύσκολα φτάνουν στη χώρα. Το ιατρικό υλικό και εξοπλισμός λείπει. Είναι απελπισμένος ο λαός της ΑΕΤ και είχε να αποθέσει όλες τις ελπίδες στην διεθνή κοινότητα. Κυρία Επίτροπε λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το πολύ απλό. Πού είναι το σύνολο τη βοήθεια που έχει υποσχεθεί στην ΑΕΤ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο η ανθρωπιστική βοήθεια. Εάν είχε φτάσει πιο γρήγορα, δεν πιστεύετε ότι αυτή τη νέα τραγωδία θα την είχαμε αποφύγει. Και πώ γίνεται για άλλη μια φορά οι διεθνεί συζητήσει να έχουν καταλήξει σε φρούδε υποσχέσει. Γιατί δεν δεν έχει προχωρήσει η επιχείρηση ανοικοδόμηση τη χώρα υπό την αγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει ο λαό τι αετή εκλογέ, αλλά υπό ποιε συνθήκε θα γίνει και με ποια στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συγγραμμένου ομιλητές. πρώτα η κυρία Ροντζούλη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρά τις εκκλήσεις για να μην ε, μειωθεί η επαγρύπνησή μας μετά τους νεκρούς του Ιανουαρίου ε, στην ΑΕΤ, οι τελευταίες ειδήσει δείχνουν τον ίσο αυτή την εγκαταλείψαμε στην τύχη της. Η διεθνής κοινότητα την εγκατέλειψε στην πιο κρίσιμη στιγμή, τη στιγμή της ανικοδόμησης. Και αυτή τη στιγμή με τις διαστάσεις που έχει πάρει η επιδημία της χολέρας γίνονται πολλά σχόλια και όλοι καταλήγουν να αποδίδουν μια μυστικιστική αξία, μια θρησκευτική αξία κιόλα στην κατάσταση της χώρας αυτής. Εάν υπήρχε ανθρωπιστική δράση δεν <coughs> δεν θα υπήρχαν ε, αυτά τα προβλήματα. Αρκεί ένας ε, στρατιώτης λόγου χάρη να προσβληθεί από τους υπεύθυνους των ξένων δυνάμεων να φτάσει στο Γενικό Επιτελείο και να μολύνει και όλους τους υπόλοιπους. Είναι πολύ μεγάλος λοιπόν ο κίνδυνος και να μην ξεχνάμε ότι μετά τα τόσα θύματα που είχαμε τον, ε, από το σεισμό του Ιανουαρίου οι άνθρωποι μένουν πλέον στις πλατείες και στους δρόμους. Αυτό φυσικά δημιουργεί συνθήκες ε, διάδοσης της ασθένειας πολύ πιο ε, κατάλληλες και έχουν αυξηθεί οι αριθμοί των νοσηλευωμένων, των ασθενών. Είναι 1130 οι προβλημένοι από την ασθένεια όπως ακούσαμε. Θα φτάσουν πολύ ψηλότερα νούμερα και ακούμε νέα ειδήσει για την εξάπλωση τη επιδημία καθημερινά. Θα πρέπει λοιπόν η διεθνή κοινότητα να πάψει να είναι αδιάφορη. Θα πρέπει αμέσω να βρούμε μια λύση. Ιδάλω, οποιοδήποτε μέρο προσβληθεί από την ασθένεια και οποιοδήποτε άνθρωπο χάσει τη ζωή του θα είναι ένα βάρο στη συνείδησή μα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον συντονισμό από τον οποίο ξεκινήσατε και τις συζητήσεις που έχετε με τη Βαρόνια Έιμο στον ΟΗΕ. Διότι το φθηνότερο πράγμα τώρα είναι να κατακρίνουμε. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να πιέσουμε αυτούς που πρέπει. Και θέλω να πω εδώ σε όλους τους ευρωβουλευτές ότι πρέπει να πιέσουμε τα κράτη μας να βοηθήσουν περισσότερο. Διότι αν δείτε τον κατάλογο των κρατών βλέπετε ότι όλες οι χώρες ε, δωρητές έχουν προβλήματα. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία ε, όλοι όμως έδωσαν. Ε, έρθετε λοιπόν όλοι σε επαφή με τις κυβερνήσεις σας να δεσμευτούν για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη βοήθεια και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ ότι δεσμεύσατε επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ διότι η πρώτη μεγάλη τραγωδία ήταν ο σεισμός και τώρα είναι η επιδημία της χολέρας. Κυρία Επίτροπε σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΤ εκτός από επίκεντρο ε, ενός μεγάλου σεισμού είναι και η χώρα που είναι πιο κακοκυβερνημένη στην ε, Λατινική Αμερική και αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα που ε, έχει το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό έλλειμμα κατά κεφαλήν ε, διεθνώς κι όμως αυτή τη στιγμή ε, το να ζουν παιδιά μέσα σε σκουπίδια και σε σκηνέ στους δρόμους, καταλαβαίνουμε σε τι μπορεί να οδηγήσει. Έτσι λοιπόν, εάν δεν προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση, με τη γραφειοκρατική μας μηχανή, με μια διοικητική κουλτούρα πολύ αδύναμη, τα κρούσματα θα αυξηθούν και η βοήθεια δεν θα φτάνει στο στόχο της. Και η διεθνής ε, κινητοποίηση πολλές φορές δεν είναι καλά συντονισμένη και δεν δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ήδη τον περασμένο Ιούνιο με την επισκέψη της κοινοβουλευτική αντιπροσωπείας είδαμε με σαφήνεια ότι η συγκέντρωση των στατοπέδων σε ακατάλληλες περιοχές και η συγκέντρωση αποβλήτων έδινε τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν επιδημίες, να αποκλειθούν επιδημίες. Να πως έφτασε η χολέρα. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της. Νομίζω ότι όχι μόνο στην ΑΕΤ πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, αλλά και μεγαλύτερη προστασία από πολιτικής άποψης σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Για λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια τραγωδία την οποία δεν αντέχουμε να συζητάμε. Όταν έπληξε ο σεισμός πέρυσι τον Ιανουάριο όλες ήρθαν Όλες οι χώρες ήρθαν να βοηθήσουν, στρατιωτικά ελικόπτερα, βαρύς μηχανικός εξοπλισμός, όλοι όμως τώρα έχουν φύγει. Και ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει, δεν υπάρχει οδικό σύστημα, δεν υπάρχει κανείς να συντονίσει τις ε, δραστηριότητες. Γιατί όλοι αυτοί που πήγαν ε, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Κλίντον κάποια μέρα εξαφανίστηκαν. Πότε θα εξαφανιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι γελίο. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητος για να εντείνουν τις προσπάθειες τους κατά τρόπον ώστε ο πληθυσμός της ΑΕΤΙΣ να μπορέσει να βοηθηθεί και ασχέτως του τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση στην ΑΙΤ είναι τραγική και υπάρχει, υπάρχουν ε, επιδημίες. Αυτό δεν είναι απρόσμενο αλλά τα πράγματα δεν προχώρησαν όσο γρήγορα προς το καλύτερο όσο θα θέλαμε. Ε, υπάρχουν δυσκολίες ε, και λόγω του σεισμού. Καλό θα ήταν να λειτουργεί σωστά το κράτος όμως αυτό δεν συμβαίνει και τώρα πρέπει γρήγορα να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διότι διαφορετικά θα υπάρξει και, και περαιτέρω βία και επιδημίες. Πρέπει οι καλύτεροι ειδικοί υγείας να επικεντρώσουν την προσοχή τους για να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα για την ΑΕΤ, να υπάρξει βοήθεια και χρηματική αλλά και στον τομέα της υγείας και να δράσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. που κάνατε και στην περίπτωση της IT αλλά και προφανώς όλα αυτά που έχετε κάνει και για το Πακιστάν και ξέρουμε ότι θα είστε παρούσα σε κάθε ανάγκη. Πραγματικά η καταστροφή είναι τεράστια. Μιλάμε για πάνω από χίλιου νεκρούς, 15.000 ε, ασθενείς και τα νούμερα συνέχεια αυξάνονται. Οι ανάγκη είναι τεράστιες και βλέπουμε ότι τα χρήματα που έχετε στη διάθεσή σας δεν φτάνουν. Γίνεται όλο και όλο πιο προφανές ότι χρειαζόμαστε πραγματικά και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ίσως και προφανώς πρώτα απ' όλα ένα φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές άλλα χρηματοδοτικά μέσα που θα μπορούν να ενισχύουν ε, τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες. Επίσης θα πρέπει να δούμε, Επίτροπε, και κλείνω με αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να μην επαναληφθεί το γεγονός να μεταφέρονται ασθένειες μέσα από ανθρώπους που δουλεύουν για τον ΟΝΟΙΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέλντερ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σήμερα το απόγευμα έφτασαν ε, κάποιε πληροφορίε, κάποια Ολλανδική οργάνωση η οποία δρά στην IT ε, πάνω από ένα χρόνο και μα έδωσαν μια ρεαλιστική εικόνα σε σχέση με το τι επικρατεί εκεί, σε σχέση με όσα ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε ένας βασικός δωρητής ε, για τη χώρα εκείνη και ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είμαστε μεγάλος δωρητής και έχουμε δεσμεύσει ε, σημαντικά κονδυλία δηλαδή για την Αιτή. Όμως πήγαν αυτά τα χρήματα εκεί. Δεν έχουν φτάσει ακόμα, δεν πήγαν και γι' αυτό και θα πρέπει να καταφέρουμε μια που κατάστην τόσο σοβαρή να φτάσουν εκεί αυτά τα χρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόληψη, νερό, θα πρέπει να πάνε η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά τα θέματα. Να δώσουμε νερό. Να τους δώσουμε πυρογνώμονες. Να τους βοηθήσουν όσον αφορά ε, τον υδροφόρο ορίζοντα και ε, γενικά υπάρχει έλλειψη όσον αφορά τα πάντα για τη χώρα εκείνη και θα πρέπει να, να λάβουν δράση οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπή Δαμανάκη, πρώτα-πρώτα θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προσπάθειε που κάνετε για την ΑΕΤ. Όμω, απαιτεί η κατάσταση αυτή τα πράγματα να γίνουν ε, πιο έντονα, πιο γρήγορα και ε, παρά το ότι έχουμε υπό την οικονομική συγκυρία κάποια δυσκολία, διότι θα πρέπει να βρεθούν τα χρήματα ε, μια που υπάρχουν για άλλε δουλειέ. από πλευράς υγεία, από πλευρά ανθρωπιστική. θα πρέπει κάτι να κάνουμε να έχουμε ε, ε, αντιμετώπιση τη ασθένεια, καθαρό νερό και όλα αυτά επήγουν. οπότε χρειάζεται να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη περισσότερο. Ο κύριος Στάκουλα για ένα λεπτό.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 Ευχαριστούμε την Επίτροπο Γιώργη για, την... για το έργο της και το έργο ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε την ΑΕΤ και να υπάρχει και προβολή της προσπαθίας μας. Αυτό είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στους πολίτες της ΑΕΤ και ότι έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας απέναντί τους. Υπέφεραν εξαιτία του σεισμού και τώρα υποφέρουν εξαιτία της επιδημίας φολέρας. Θα πρέπει λοιπόν όταν προγραμματίζουμε να αποστείλουμε κονδύλια αυτά να φτάνουν εγκαίρως οι, βοήθη, οι οργανώσεις ε, για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια έχουν κάνει εξαιρετικό έργο και έχουν ανοίξει τους διάβλους που χρειάζονται ώστε να φτάνει η βοήθεια σε αυτούς που την ε, έχουν περισσότερο ανάγκη. Ελπίζω λοιπόν ότι της του μηχανισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας ή τις χριστιανικές οργανώσεις θα τις αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε στην πράξη να μπορέσουν να λάβουν δράση και να είμαστε βέβαιοι ότι τη βοήθεια θα την στείλουμε στους ανθρώπους αυτούς ώστε να συντομότερα για να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας και τη συζήτηση ενός θέματος το οποίο ατυχώς θα παραμείνει επί αρκετό καιρό διότι δεν είναι μια εύκολη κρίση για να επιληθεί. Είχαμε ορισμένους, κάνει ορισμένους υπολογισμούς σχετικά με την κλίμακα του προβλήματος για τους επόμενους μήνες προτού εξελιχθεί και αναφέρομαι στους δικούς μας εμπειρογνώμονες και συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι πρέπει να στείλουμε εμπειρογνώμονες ε, στην ΑΕΤ διότι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου των Καταστροφών μας λέγουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μολυσμένοι με το, την ασθένεια και ε, το, στο ίδιο υπολογισμό 400.000 ε, καταλήγει και η Παναμερικανική οργάνωση γι' αυτό και συμφωνώ αμέσως πρέπει να κινητοποιηθούμε πρέπει να βοηθήσουμε αμέσως και θέλω να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία καταρχήν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα είναι μια στιγμή όπου θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε τις οργανώσεις που είναι εκεί να να τους δώσουμε τους πόρους για να ενεργήσουν και συγχρόνως θα πρέπει να βοηθήσουμε διότι όταν αναφέρομαι στα κράτη-μέλη μιλώ σαν να μιλώ σε αδέρφια μου διότι πιστεύω ότι κάνουμε μεν αλλά χρειάζονται πολλά παραπάνω από το υγειονομικό προσωπικό από δισκία για να καθαρίσει το πόσιμο είδωρ. Πολλοί εδώ μίλησαν ε, για την τεράστια παρανόηση του τι είναι αυτή η ασθένεια και πώς μπορεί ε, καλύτερα να ε, αντιμετωπιστεί και πολλοί πεθαίνουν διότι δεν πηγαίνουν στους υγειονομικούς σταθμούς γιατί φοβούνται ότι θα μολυνθούν και όχι ότι θα τους γιατρέψουν. Επίσης πολλοί μίλησαν για τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί να δώσουν οι δωρητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τιμήσει την υπογραφή της, δώσαμε τα 60 εκατομμύρια με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε καθορίσει. Είπατε ε, ε, ε, η Κάθη Άστον και ο Επίτροπος Πίμπαλς θα κοιτάξουν με τα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε ένα απολογισμό για το τι έγινε με τα χρήματα τα οποία δώσαμε και αυτό είναι πολύ σοβαρό διότι η φήμη της διεθνούς κοινότητος διεκυδεύεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και έρχομαι σε ένα πολύ βασικό θέμα υπάρχει ε, ε, ένα όριο στη δυνατότητα αφομοιώσεως ε, στην IT και αντιλαμβάνομαι ότι θα με καταλάβατε αν πω ότι όταν πρωτοπήγα στην Αιτή είπα ότι ίσως δεν ήταν το χειρότερο πρόβλημα της ΑΕΤ. Το χειρότερο πρόβλημα στην Αιτή είναι ότι επί δεκάδες χρόνια δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος και υπάρχει έλλειψη αναπτύξεως οπότε δεν υπάρχει σωστό υγειονομικό σύστημα. Είδα στους καταβλισμούς τα παιδιά ε, ε, τα οποία φοβούνται φοβόντουσαν τον γιατρό διότι πρώτη φορά βλέπανε γιατρό στα μάτια τους και ε, ε, φοβόντουσαν τα άτομα που πήγαν να τους βοηθήσουν στους καταβλισμούς. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές δυνατότητες και δεξιότητες ενός ορθά λειτουργούντος κράτους που δεν υπάρχουν. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση ακόμη με τη βοήθειά μας να επιτρέψει να υπάρξει ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων προς αποφυγή της επεκτάσεως της επιδημίας για να βελτιωθεί η υγειονομική κατάσταση. Τονίζω λοιπόν ότι τα προβλήματα της ΑΕΤΙΣ δεν θα λυθούν απλώς διότι κατά βάθο υπάρχουν δεκάδες χρόνια με έλλειψη ανάπτυξης χωρίς ένα κράτος που λειτουργεί ομαλά και οι αρχές ε, προσπαθούν να σέβονται το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθορίσει ε, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή τη στιγμή αλλά πιστεύω ότι εάν ε, καθυστερήσουμε ή καταργήσουμε τις επερχόμενες εκλογές θα αποσταθεροποιήσουμε τη χώρα και γι' αυτό από αυτά που έχω ακούσει τουλάχιστον και όχι από ό,τι έχω δω αυτή είναι η γνώμη που έχω διαμορφώσει. Το τέταρτο θέμα μου είναι η εμπλοκή που με ζητήσατε μα είπατε να εμπλακούμε άμεσα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το πράξουμε. Η Βαρόνια, Άμος αύριο θα είναι ήδη στην ΑΕΤ και θα πάω και εγώ διότι αυτή τη στιγμή η κινητοποίηση, ο καλός συντονισμός και ειλικρινά το να δώσει κανείς ελπίδα στους ανθρώπους εκεί και στο προσωπικό μας το οποίο παλεύει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση σε περιοχές όπου η γεωνομική ε, υπεύθυνη στην ΑΕΤ ε, εγκαταλείπουν και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την τεράστια αύξηση των ασθενών. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε μία ψύχρεμη παρεσία και ε, να προσπαθήσουμε να ε, δώσουμε ελπίδα στο λαό. Ένας ομιλητής είπε ότι είναι ανθεκτική η κάτοικη της ΑΕΤΙΣ. Όντως και αυτή είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Η συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία.